Είναι σαφές λοιπόν γιατί η Δανία θέλει να παραμείνει εκτός της Ευρωζώνης. Θέλουμε να ασκούμε τη δική μας οικονομική πολιτική. Δεν είναι θέμα άλλων εθνικότητων αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. 7 Απριλίου, τη Δετάρτη, στη 2.30 επαναλαμβάνεται η σύνοδος, η δική σύνοδος για την εξέταση των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Συνόδου. Λύεται η συνεδρίαση.